Ε, τα... Τα πρακτικά συνεδρία θα υποβληθούν στην αρχή της επόμενης ε, συνεδρίασης. Στο Κοινοβούλιο δεν έχετε άλλες παρατηρήσεις. Τα ψηφίσματα που υιοθετήσαμε στη σημερινή συνεδρίαση θα προωθηθούν στα αρμόδια σώματα που αναφέρονται στα ίδια τα ψηφίσματα.